ενδιαφέρον εργάστηκα με τους συναδέλφους και χαίρομαι που ο συμβιβασμός αυτός ε, τήρει την, ε, την ψηφοφορία που είχαμε, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Φαντάζεστε την απογοήτευση του Πρόεδρου σας που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε αυτή την συζήτηση. Γι' αυτό ο Πρόεδρος σας εκμεταλλεύεται το δικαίωμα που έχει να συγχαρεί την κυρία Τράπτμαν, την κυρία Ντελκαστήγιο και ε, την κυρία, τον κύριο συγγνώμη Χάρμπορ ε, για το έργο τους και ιδιαίτερα την ε, Επίτροπο Ρέντινγκ με την οποία συνεργάστηκαν και οι τρεις εισηγητές θαυμαστά. Θα ήταν μεγάλη χαρά μας να φιλοξενήσουμε και το Συμβούλιο εδώ. Και έτσι θα είχαμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε και ε, ορισμένες νομικές πτυχές των ε, κάπως ε, περίεργων αυτών επιστολών του Συμβουλίου. Και προχωρούμε τώρα στην κοινή συζήτηση για την Europol. Δεν ξέρω αν είναι παρόν ο κύριος Νίκολσον. Είναι. Here. Okay. Οπότε τον λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Νίκολσον, για τέσσερα λεπτά. Mr. Nicholson, you have the floor for four minutes. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό το timing. Μια φορά στη ζωή μου. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Κέρκοπ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί. Οπότε θα διαβάσω τα σοφά λόγια τα οποία έγραψε και μου ενεχείρισε για να σας διαβάσω. Εις ό,τι αφορά την προσαρμογή των κανόνων για την εμπιστευτικότητα των ε, πληροφοριών της Europol. Οι κανόνες που θα πρέπει να υιοθετηθούν θα αντικαταστήσουν μέτρα ασφαλείας για όλες τις πληροφορίες που επεξεργάζεται η Europol. Με άλλα λόγια, ένα κοινό πρότυπο για την προστασία των πληροφοριών που περνούν από ε, τους διάβλους, από επικοινωνίας ε, μεταξύ Ευρωπόλ και κρατών μελών. Η διαπραγμάτευση του χρονοδιαγράμματος ήταν ε, οδυνηρή διαδικασία με την υπογραφή της συνθήκης της ε, Λισαβόνας, την επικύρωσή της καλύτερα, οι διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή ΛΑΝΚΕ είναι πλέον ξεπερασμένες. Υπάρχει και μια άλλη επιτροπή, ε, έκθεση που ζητεί από τους συναδέλφους να απορρίψουν το κείμενο του Συμβουλίου. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι υποστηρίζουμε τον στόχο του Συμβουλίου γιατί υποστηρίζουμε την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και αναγνωρίζουμε τα ωφέλη της Europol στην καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του πολίτη. Η υπηρεσία θα πρέπει να είναι ώστε να τον πιο αποτελεσματική και βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και την κυριαρχία των κρατών μελών εις ό,τι αφορά την, ε, τον έλεγχο των αστυνομικών τους δυνάμεων. Υποστηρίζουμε βέβαια την Ευρωπαϊκή Αστυνομία με την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας και αυτό θα επηρεάσει την αστυνομική συνεργασία. Ο εισηγητής πιστεύει και οι συνεισηγητές του στην Επιτροπή ΛΥΒΕ πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στην απόφαση η Europol μέχρι τέτοιου είδου μέτρα να μπορέσουν να υιοθετηθούν δυνάμει του νέου νομοθετικού πλαισίου που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνα. Καλούμε λοιπόν το Συμβουλίο. Καλούμε λοιπόν το Συμβουλίο, διακόπτει ο Πρόεδρος. Μπορείτε να επιβραδύνετε κύριε Νίκολσον. Μα αλίμονο, Πρόεδρε, αλίμονο. Με τα χαράς να επιβραδύνω Ζητώ συγγνώμη. Έλεγα ότι ο εισηγητής καλεί το Συμβούλιο να αποσύρει την πρότασή της και να κάνει μια δήλωση στην Ολομέλεια επί της δηλώσεως για μια νέα απόφαση της Europol που θα υποβληθεί έξι μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνος. Τώρα θα ήθελα να στραφώ στην δεύτερη έκθεση πρωτοβουλία της Ισπανίας και της Σουηδίας για μια οδηγία για τις εργαστηριακές δραστηριότητες της Europol. Η, το βασίλειο της Ισπανίας και το βασίλειο της Σουηδίας θέλουν συμβεβλημένα εργαστήρια να μπορέσουν να συνεργάζονται με την Europol και αυτό προ όφελο τη καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών τα τελευταία χρόνια. Η ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα αυτό τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία είναι υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή στα πλαίσια τη προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος γενικότερα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών διαδικασιών σε ένα κράτος μέλο θα αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό προ χάρη τη νομική ασφάλεια, τους υπόπτου, αλλά και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Οι εργαστηριακες, λοιπόν διαδικασίες θα πρέπει να είναι συμβεβλημένες για το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα των εργαστηρικών του δραστηριοτήτων αναγνωρίζονται στα άλλα κράτη-μέλη ως ισοδύναμα των ιδίων των συμβεβλημένων του εργαστηρίων. Βεβαίω η ίστατη ε, αρμοδιότητα είναι στα χέρια της εκάστοτε δικαστική αρχής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας. Έχω μία ακόμα παράγραφο να διαβάσω, Πρόεδρε, και συγγνώμη αν τα λέω πάλι γρήγορα. Η νομική βάση αποτελεί ένα πρόβλημα, αλλά με την συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε πλέον τη δυνατότητα να απορρίψουμε την πρωτοβουλία του Βασιλείου της Ισπανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τη νέα νομική βάση, επί τη βάση της νέας νομικής πραγματικότητας. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να εξετάσουμε με περισσότερο χρόνο και σε μεγαλύτερο βάθος το θέμα αυτό, διότι ο χρόνος πίεζε μέχρι τώρα και δεν είχαμε δυνατότητα να το πράξουμε ως θα έπρεπε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη που μιλώ ογκρικά. Ανέλαβα εγώ την Προεδρία. Δώσαμε την ευκαιρία στον κύριο Νίκολσον να μιλήσει λίγο παραπάνω, γιατί έτσι μιλούσε και λίγο πιο αργά. Το λόγο έχει η κυρία τη Σοφή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη εγώ και ίσως να αντισταθμίσω έτσι το χρόνο του κυρίου Νίκολσον. Για να μην ε, ε, έχουμε και υπέρβαση. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνθήκη της Αβώνας θα δεθεί σε ισχύ σε 7 ημέρες και 5 ώρες από τώρα, αν είμαι σωστή στους υπολογισμούς μας. Και πρέπει να σας πω ότι το Συμβούλιο βιάζεται να πάρει κάποιες αποφάσεις και αυτό είναι κάπως ενοχλητικό και μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Επίσης ενοχλητικό είναι το άδειο έδρανο εδώ. Ε, θα ήλπιζα να δω παρόν το Συμβούλιο για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων αν μη τι άλλο. Ουσιαστικά συμφωνούμε με τις προτάσεις του προηγούμενου ομιλητή. Βεβαίως υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της Europol. Θέλουμε ισχυρή Europol, θέλουμε ε, μια υπηρεσία που να μπορεί να λειτουργεί σωστά και να εγγυάται ε, την ελευθερία μας και να καταπόλεμα το έγκλημα, αλλά να υπόκειται και σε δημοκρατικό έλεγχο. Γι' αυτό δανείζομαι την ε, πρόταση του προαλήσεδες και συμφωνώ και καλώ το Συμβούλιο να αποσύρει τις προτάσεις για το Europol και να καταθέσει νέα πρόταση το αργότερο εντό 6 μηνών και κατά προτίμηση νωρίτερα υπό τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και τέλο, για το τελευταίο, το ειδικό θέμα που με αφορά εμένα και η μισηγήτρια για τη ε, διαβίβαση εμπιστευτικών εγγράφων και προσωπικών δεδομένων σε τρίτεους θα ήθελα να ακούσω το Συμβούλιο που απουσιάζει κατά τα άλλα να μα πει ε, πώς εκλαμβάνει την ανάλυση ε, της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φρονεί ότι η νομική βάση που έχετε επιλέξει είναι λάθος. Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου. Μήπως ε, επανέλθουν κάποια στιγμή, ε, βρουν κάποιον να μπορέσει να μας δώσει καμία απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιάνν Φιλίπ Άλμπερτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Er ε, είναι πολύ καλό αυτό που είπαν οι πρόεδροι και θα ήταν συνεπές και μόνο να αποσύρει ε, την πρόταση του συμβουλίου και να φέρει νέα πρόταση για την Europol υπό τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Είναι σωστό και χρήσιμο η δικαστική και αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη να ελέγχεται και να συζητήσει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρχει και συναπόφαση. Μόνο έτσι μπορεί η εργασία τη Ευρωπόλ να προχωρήσει και να έχει και απαραίτητη και αρκετή νομιμοποίηση. Μόνο αν από κοινού ενωμένοι ε, αποκρούσουμε και ε, την πρόταση του Συμβουλίου και την αποσύρει, θα καταλάβει το Συμβούλιο περί τίνος πρόκειται. Χρειάζεται αλλαγή και η νομική βάση. Κατά τα άλλα υπάρχει και ο εξής λόγος. Επί ε, πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό όλα αυτά τα αποφάσισαν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους διακυβερνητικά. Εγκρυπτό και παραβίστο. Το αργότερο στις 11 Σεπτεμβρίου έχουν ε, αποφασίσει πακέτα ασφαλείας που η αποτελεσματικότητά τους, η αναλογικότητά τους και η σκοπιμότητά τους δεν έχουν ε, εγκριθεί ούτε καν ελεγχθεί ούτε καν συζητηθεί ποτέ. Τρίτος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους επέτρεπε να αποφασίζουν οι κυβερνήσεις και να παρεμβαίνουν με τρόπο πάρα πολύ αμφιλεγόμενο στις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. Και υπάρχει μια επικίνδυνη ανισορροπία αυτή τη στιγμή. Η συνεργασία των αρχών ασφαλείας παγκοσμίω στενεύει όλο και περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα η Διεθνή Συμφωνία για ελάχιστε προδιαγραφές για προστασία των δικαιωμάτων απουσιάζει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, το χάσμα αυτό διευρύνεται μεταξύ των κρατικών εξουσιών και των δικαιωμάτων των πολιτών. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Ασφαλείας Europol, Eurojust και Frontex και το σύστημα πληροφορία Schengen, Eurodat και πάει λέγοντας, όλο και περισσότερα στοιχεία δεδομένα ε, συλλέγονται, συσσωρεύονται, ε, ε, προχωράει η αξιοποίησή τους και η ανταλλαγή πληροφοριών και στην Ευρώπη γίνεται όλο αυτό το σύστημα και πιο θολό. Δεν ξέρουμε ποιος χρησιμοποιεί ποια δεδομένα και μπορεί να τα συλλέγει, να τα κατέχει, να τα αξιοποιεί, να τα εκμεταλλεύεται, να τα διαβιβάζει. Υπολείπεται κατά πολύ ο έλεγχος. Και τι θα γίνει αν όλα αυτά τα στοιχεία τα δίνουμε σε τρίτες χώρες. Και δεν πρόκειται πάντα για την Ορβηγία, για τη Σουηδία για την Ελβετία. Έχουμε και η παρουσία, μέχρι και Μαρόκο και Κίνα πάει η ιστορία αυτή. Ερωτώ, ποιος μπορεί να εγγυηθεί προστασία από την κρατική αυθαιρεσία. Όχι, το Κοινοβούλιο όχι. Το Κοινοβούλιο έχει και την ε, εξουσία και το καθήκον, αλλά έχει και την αξίωση να συμμετέχει στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και στη διεθνή συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της ε, τρομοκρατίας, χωρίς κανένα περιορισμό των δικαιωμάτων. Αυτή η δημιουργία κοινών ελαχίστων προδιαγραφών και προτύπων θα πρέπει να γίνει πριν προχωρήσουμε στη σύναψη περαιτέρω συμφωνιών για ανταλλαγή στοιχείων με τρίτες χώρες. Αυτό ισχύει και για τις πληροφορίες της Europol αλλά και για τα SWIFT στις τράπεζες, για τα ε, δεδομένα των επιβατών που ανταλλάσσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σαφή πρότυπα για την προστασία, ε, έλεγχος σκοπιμότητας και αναλογικότητας και προστασία των πολιτών είναι το πρώτο βήμα και απαραίτητη προϋπόθεση. Χαίρομαι που στο πακέτο ε, για την Ευρωπόλ συμφωνούμε πέρα από πολιτικές ομάδες και το θεωρώ και καλό σημάδι για την επικείμενη συζήτηση για μια ευρεία προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλμπρέχτ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δίας Δεμέρα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πακέτο Europol αποτελείται από τέσσερα σχέδια απόφασης που στόχο έχουν την ανάπτυξη, του, την εφαρμογή του, της απόφασης του Συμβουλίου του Απριλίου του 2009. ζητώ και εγώ, όπως άλλοι συναδελφοί, την απόσυρση της πρότασης του Συμβουλίου. Θέλουμε το Κοινοβούλιο να έχει πολύ πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και η συνθήκη της Λισαβόνας να είναι η νομική βάση για την απόφαση Europol. Θέλουμε το Κοινοβούλιο και το Συνομβούλιο να είναι σε ισότιμη και ισορροπημένη θέση. Για να κατανοήσετε καλύτερα τους λόγους της απορριψής μου θα πω δύο λόγια για το αντικείμενο της έκθεσής μου. Μία από τις βασικές αρμοδιότητες της Europol είναι η αποθήκευση, η επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων. Για να αναλυφθεί αυτό το σημαντικό έργο πρέπει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να δίδουν πλήρες πληροφορίες στην Ευρωπόλ, ενημερωμένες και ακριβείς. Μόνο έτσι η Ευρωπόλ θα μπορέσει να έχει το αναλυτικό έργο που θέλουμε να έχει. Στα πλαίσια της απόφασης του Συμβουλίου, στο άρθρο 2, αναφέρονται και δεδομένα προς ε, ανάλυση, σύμφωνα με την εντολή που υπάρχει στο άρθρο 14.1. Έτσι, η Ευρωπόλ έχει 19 αρχεία διαφορετικά. Κάθε αρχείο είναι μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων που διασυνδέεται με τις άλλες και που συνδέεται από μόνο του με μια συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα και κάθε αρχείο συνδέεται με τη συγκεκριμένη μορφή υποστήριξης που μπορεί να παράσχει η Ευρωπόλ. Τα αναλυτικά αυτά αρχεία σήμερα είναι το μόνο νομικό εργαλείο που έχει η Ευρωπόλ για να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί και να αναλύσει δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών. Επίσης υπάρχουν γενικές αρχές και κανόνες τόσο τεχνικής φύσεως όσο και κανόνων χρήσης αυτών των στοιχείων. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να έχουμε ένα νομικό μέσο που θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπογραμμίζω, τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και επίσης την πλήρη ε, ανάληψη των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Ευρωπόλ. Σε αυτά τα πλαίσια ερωτώ, είναι σωστή ή όχι η νομική βάση που προτίθεμεθα να εφαρμόσουμε. Ως προς αυτό, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως σώμα εκπροσώπησης των πολιτών είναι απαρέγκλητος και απαρέγκλητος είναι και ο έλεγχος που θα πρέπει να ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο λοιπόν εν ώψη τη άμεση θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην νομοθετική διαδικασία σε ισότιμη βάση με το Συμβουλίο. Κανένα κριτήριο επίγοντο χαρακτήρα δεν μπορεί να καταστρατηγήσει την αρχή αυτή. Ζητώ λοιπόν από τους αξιότιμους συναδέλφους να μας υποστηρίξουν, να υποστηρίξουμε δηλαδή την ε, υπηρεσία της Ευρωπόλ αλλά προς το παρόν να απορρίψουμε την του Συμβουλίου μέχρι να στηριχθούμε στη νέα νομική βάση που προσφέρει συνθήκη της Λισαβόνας. Ζητούμε από το Συμβούλιο να αποσύρει την πρόταση και να παρουσιάσει μια νέα σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Κύριε Πρόεδρε, σε άλλο γύρο τραπέζης θα προβώ σε πιο βαθίες και επεξηγηματικότερες διευκρινήσει τη θέσεώς μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διεσδεμέρα. Επόμενη ομιλήτρια τώρα είναι η κυρία Σόνια Αλφάνο. Για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε για το δίκτυο πρόληψη του εγκλήματο. Δημιουργήθηκε το 2001 με απόφαση του Συμβουλίου 2001 κάθετο η στόχη αυτού του δικτύου είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας, η ανταλλαγή πληροφοριών και της, ε, των εμπειριών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών, η οργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων, πρωτοβουλειών που έχουν ως στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και βελτιστών πρακτικών, και βεβαίω ε, παροχή πληροφοριών και συμβουλών προ το Συμβούλιο, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόληψη του εγκλήματο. Είπε αρχικά η δομή αυτή να βασιστεί σε σημεία επαφή τα οποία διορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Έναν εκπρόσωπο ανά αρχή και άλλα ε, σημεία επαφή τα οποία θα μπορούσαν να διοριστούν μεταξύ του ερευνητών ή καθηγητών ε, πανεπιστημίων, εξειδικευμένων κτλ. Τα κράτη-μέλη παρόλα αυτά έχουν υποχρέωση να δώσουν δυνατότητα ε, συμμετοχή ΜΚΟ τη Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών και του ακαδημικού κόσμου. Το παρατηρητήριο τη Λισαβόνα επίση συμμετείχε. Το 2005 το δίκτυο υπευλήθη σε μια πρώτη εσωτερική μεταρρύθμιση. Δημιουργήθηκαν δύο επιτροπές, η μία για το πρόγραμμα εργασίας και η άλλη για την έρευνα. Ενώ η, το, η σελίδα ε, πέρασε σε αρμοδιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2007 έγινε μια νέα μεταρρύθμιση που στόχο είχε την ενίσχυση της γραμματείας. Και βεβαίω, έθεσε και θέμα πόρων των μονιμών αντιπροσωπιών. Χρηματικό δηλαδή, δημοσιονομικό. Το Μάρτιο του 2000. ανατέθηκε και δημοσιεύτηκε σε, από σύμβουλο μια έρευνα για τους λόγους στους οποίους οδηγήθηκε σε αποτυχία οργανωτική η υπηρεσία αυτή και που βεβαίως σε δυνατότητα στην επιτύχει του στόχου της. Το δίκτυο δηλαδή έλλειψη ίδιων πόρων, αναποτελεσματική γραμματεία, μη συμμετοχή των εθνικών εκπροσώπων και πολύ πτωχό πρόγραμμα εργασίας. Επίσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση, υποβλήθηκε και η πρόταση να διαλυθεί το δίκτυο. Συστάθηκε ομάδα εργασίας για να εξετάσει τις, προσ... τις ε, προτάσεις αυτές. Και αποφάσισε ότι θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό του δικτύου εξωτερική γραμματεία προτάθηκε με χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια, από κονδύλια από κοινοτικά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, ε, παρόλο που ορισμένα κράτη-μέλη δεν ήθελαν να. μάλλον δέχτηκαν τη διάλυση του δικτύου, άλλα κράτη-μέλη δέχτηκαν τη μεταρρύθμιση αυτού. Και η Προεδρία του Συμβουλίου, η Σουηδική Προεδρία, υιοθέτησε αυτή την πρόταση Δηλαδή να καταστήσει προτεραιότητα ε, το θέμα αυτό στα πλαίσια του προγραμματός της. Ως εκ τούτου και εγώ εκφράζω την λύπη μου, την αμηχανία μου για τον κενό θόκο, για την απουσία εκπροσώπου του Συμβουλίου, της Προεδρίας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθε στο εμπαρόδο αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν δημιουργήθηκε και το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από, εθνικούς, από εθνικά μέλη που ορίζουν τα κρατη και το οποίο θα προεδρεύει ένα πρόεδρο επικεφαλή εκτελεστική επιτροπή. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια σύγχυση εδώ μεταξύ των σημείων επαφή των εθνικών αντιπροσωπιών. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό διότι, διότι λέγω, διότι δεν συμμετέχει πλέον η, κοινο... η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, ο ακαδημαϊκός κόσμος, οι εμπειρογνώμονες, οι ερευνητές. δεν συνδέεται καθόλου το δίκτυο με τα άλλα κοινοτικά όργανα που ασχολούνται με το θέμα του εγκλήματος και της προλήψεως αυτού. Δεν προβλέπεται καμία δε μορφή συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καταστρατηγείται εντελώ η προϋπόθεση γνώσεις ξένων γλωσσών, που είναι απολύτως απαραίτητη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν επέτευσαν οι στόχοι για του οποίου δημιουργήθηκε το δίκτυο. Δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ κομισιών, κρατών μελών, συμβουλίου. Θα το έλεγα δράση σαμποτάζ κατά του ιδίου του δικτύου δολιοφθορά κατά του ιδίου του δικτύου. Οι εμπειρογνώμονες που ήταν σε επίσκεψη σε άλλη χώρα δεν μπορούσαν πολλές φορές για να μην πω πάντα να συνεννοηθούν διότι δεν προβλέπεται μετάφρασης. Κάτι το οποίο καθιστά εντελώς αναποτελεσματικό το δίκτυο. Ευχαριστώ. Πρέπει να ενδυναμώσουμε λοιπόν την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος από, με όλες τις δυνατότητες που έχουμε και προς τούτο το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, αναγνωρίσει ότι είχε με μια φιλόδοξη πρόταση την οποία όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριο Ζακ Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον τι διάφορε παρεμβάσει του κυρίου Νίκολσον, της κυρία Τινβέλτ, του κυρίου Άλμπρεχτα και της κυρίας Αλφάνο. Βεβαίως είναι μια συζήτηση όπου έχουμε τα διαδικαστικά προβλήματα και τα προβλήματα ουσίας μορφής και ουσίας. Για τα προβλήματα τα διαδικαστικά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε την παραμονή της θέσης σε ισχύ του συνθήκης της Λισαβόνας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα ερωτηματικά τα οποία μπορεί να προκαλέσει στο Κοινοβούλιο η έγκριση από το Συμβούλιο ορισμένων αποφάσεων. Είναι αληθές ότι η Κομισιόν λυπάται για αυτή την κατάσταση κάπως, αλλά θα ήθελα να σας διαφωτίσω λίγο για αυτούς τους τρεις φακέλους εδώ στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπόλ, όπως γνωρίζετε, με μια απόφαση του Συμβουλίου θα αντικαταστήσει την διακυβερνητική σύμβαση και θα έχει ένα νέο νομικό πλαίσιο και θα γίνει την 1η Ιανουαρίου του 2010 μια υπηρεσία, μια υπηρεσία της Ευρώπης. Όπως ξέρετε, μακρές διαπραγματεύσεις προηγήθηκαν της λήψης αυτής της απόφασης του Συμβουλίου και οι προετοιμασίες για την υλοποίηση της απόφασης λαμβάνουν χώρα τώρα. Καταλαβαίνω πολύ καλά τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και συμμερίζομαι τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου ότι περιμένει να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο το θεσμικό διότι αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ανοίξει το δρόμο για έναν έλεγχο δημοκρατικό πληρέστερο για τον ε, Ευρωπαϊκό Γραφείο Αστυνομίας. Και θα πρέπει και εμείς να εξαγάγουμε συμπεράσματα και διδάγματα από αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου για να έχουμε μια στερεά βάση για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε την μελλοντική μας νομοθεσία. Και γι' αυτό βεβαίως θα είναι ενδιαφέρον να συνδέσουμε το Κοινοβούλιο όπως και άλλα εμπλεκόμενα μέρη στην επόμενη ρύθμιση του θέματος της Ευρωπόλ. Και κυρίως για τον τρόπο άσκησης του ελέγχου από το Κοινοβούλιο και από, τις εθνική τα εθνικά κοινοβούλια ε, των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Αυτά κύριε Πρόεδρε είχα να πω, αλλά παρόλα αυτά λυπούμε που το Κοινοβούλιο απορρίπτει τα σχέδια αποφάσεων του Συμβουλίου. Πρόκειται για διατάξεις υλοποίησης εφαρμογής, εφαρμοστικές διατάξεις που θα ρυθμίζουν ε, σημαντικές απόψεις της δραστηριότητας της Ευρωπόλ, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει η Ευρωπόλ. Έρχομαι τώρα στις, τα εργαστήρια τα επιστημονικά της αστυνομίας και εδώ καταλαβαίνω που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε μια άλλη βάση για αυτήν την απόφαση πλαίσιο σχετικά με την διαπίστευση των δραστηριοτήτων των ανακριτικών ε, εργαστηρίων της αστυνομίας. Εμείς είμαστε στην Κομισιό υπέρ της διαπίστευσης, διότι έτσι θα προωθήσουμε την ποιότητα της εργασίας αυτών των εργαστηρίων, κυρίως όσον αφορά στις ευαίσθητες τεχνικές που σχετίζονται με τα δακτυλικά αποτυπώματα, με τα δείγματα IDN, DNA και όσο περισσότερο θα έχουμε διαπιστεύσει αυτά τα εργαστηρία, τόσο περισσότερο θα είναι μεγάλη η εμπιστοσύνη των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών. Καταλαβαίνω πολύ καλά άλλη μια φορά το πρόβλημα της νομικής βάσης. Η Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο, είναι της άποψης ότι η απόφαση πλαίσιο εφόσον αναφέρεται σε υπηρεσίες με την έννοια του άρθρου 50 της συνθήκης που θέσπισε την ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει ε, να έχει αυτό το άρθρο 50 ως νομική βάση. Και έτσι η... στην Κομισιόν κάναμε μια δήλωση εξ ονόματος της Κομισιόν ε, που βρίσκεται στα πρακτικά της Συμβουλίου Τζάι της 23 Οκτωβρίου 2009 και στη δήλωση αυτή η Κομισιόν βεβαίως επιφυλάσσεται το δικαίωμα να λάβει στο μέλλον τα μέτρα που θα κρίνει απαραίτητα. Προσθέτω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του οικονομικού κανονισμού, η Κομισιό είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των 100 μελών που θα επιτρέψουν την διαπίστευση ε, των εργαστηρίων της, ε, των επιστημονικών της αστυνομίας. Τέλος, η Κομισιό είναι διατεθειμένη να προβεί σε μια αξιολόγηση της υλοποίησης και της εφαρμογής του μέσου αυτού την πρώτη, για την 1η Ιουλίου 2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.4 νέο. Σχετικά με τη διαπίστευση αυτή καταλαβαίνω πολύ καλά τη θέση του Κοινοβουλίου αλλά είμαι της άποψης ότι κατά βάθο η διαπίστευση αυτή ε, είναι ε, ορφή και βάση των επιθυμιών που εκφράστηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο. Έρχομαι τώρα στην European Union Crime Prevention Network στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πρόληψη της εγκληματικότητας. Η, ε, η δίωξη δεν αρκεί. Για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε το ε, οργανωμένο έγκλημα και την παραβατικότητα, είτε πρόκειται σε εθνικό επίπεδο είτε σε διασυνοριακό, η πρόληψη είναι απαραίτητη και εξάλλου στις πρόσφατες προτάσεις τις οποίες έκανα ε, σχετικά με το εμπόριο των ανθρώπων, σχετικά με την παιδοπορνογραφία ε, ε, πρότεινα μέτρα προληπτικά. Η κυρία, κυρία Αλφάνο δείξατε τις αδυναμίες του δικτύου. Αναφερθήκατε σε αυτές. Είναι αλήθεια ότι μια πρόσφατη αξιολόγηση κατέληξε ότι οι ανάγκες της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι πραγματικές για την πρόληψη της, του οργανωμένου εγκλήματος και είναι αληθές επίσης ότι οι δημόσιοι οργανισμοί, οι ενώσεις, οι ιδιώτες επιθυμούν μια πολυκλαδική, πολυτομεακή προσέγγιση ούτως ώστε να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και μέσων. Είναι αληθές λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος προσέκρουσε σε δυσκολίες στρατηγικής φύσης, πολιτικής φύσης, ε, οργανωτικής φύσης. Η Κομισιό το συνειδητοποίησε αυτό. Αυτό που κάναμε αμέσως είναι να αυξήσουμε την, στήριξη, την οικονομική στη γραμματεία του δικτύου. Βεβαίως, στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης εμείς θέσαμε ως προτεραιότητα την αστυνομική συνεργασία και δώσαμε προτεραιότητα επίσης την αναγκαιότητα εφ' να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τρόπο ε, κοινοτικό αυτήν την ε, αστυνομική συνεργασία δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Είναι αληθές ότι το δίκτυο μπορεί και αναφέρατε ορισμένες δραστηριότητες που θα μπορούσε να επιτελέσει αυτό το δίκτυο και προτείνατε παραδείγματα ενδιαφέροντα εργασιών που θα μπορούσε να αναλάβει το δίκτυο αυτό. Μπορεί κανείς επίσης να σκεφτεί ότι κοινά προγράμματα, κοινά σχέδια θα μπορούσαν να υπάρξουν ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές, με τα σχολεία, με την ε, συνεχιζόμενη ε, εκπαίδευση, με τα προγράμματα τα σχολικά. Βρισκόμαστε στην απαρχή μιας μεγάλης πολιτικής πρόληψης της εγκληματικότητας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και του Κοινοβουλίου πρέπει να αυξηθούν, να ενισχυθούν και γι' αυτό η αστυνομική συνεργασία είναι εμπίπτη τώρα στον τομέα της συναπόφασης. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τρόπο όσο το δυνατόν στενότερο με βάση τη νέα νομική βάση και αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών που θίγονται από προβλήματα ασφαλείας στην καθημερινή ζωή. Αυτές είναι οι απαντήσεις βεβαίως. Λυπούμε κάπως για αυτή τη συζήτηση που αναφέρεται και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και στην ουσία. Αλλά πιστεύω ότι εφ' εξής, με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα της Λισαβόνας θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη δράση μας και το Κοινοβούλιο θα λάβει τη θέση που του ανήκει μέσα σε αυτή τη νέα στρατηγική κατά της οργανωμένης εγκληματικότητας και κάθε μορφής εγκληματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαρό. Ακολουθούν τώρα οι ομιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Βάντεν Κάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απαντήσεις που μας έδωσε και την περιγραφή και ε, τις εξηγήσει για τα διάφορα θέματα. Η δικαστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν μιλούμε για την Ευρώπη των πολιτών, κυρίως πρόκειται και για την ε, ε, δικαστική συνεργασία. Μέσα σε αυτή τώρα, η καταπολέμηση εγκληματικότητας είναι η πρώτη προτεραιότητα. Κυρίως επειδή η εγκληματικότητα είναι όλο και πιο διεθνής και δεν γνωρίζει σύνορα Δεν υπάρχει πλέον περιορισμένη σε κράτος μέλος εγκληματικότητα. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι μεγάλος υποστηρικτής μιας ισχυρής Ευρωπόλ και μιας ισχυρής Ευρωντάκ. Και επίσης για τα εργαστήρια ανακριτικής. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι ο δημοκρατικός έλεγχος εκείνων που καταπολεμούν την εγκληματικότητα. Δεν θέλω να το κρύψω καθόλου, αλλά να ζητήσω την προσοχή σας και για τις προτάσεις που θα έρθουν τους επόμενους μήνες για τη θέση των θυμάτων. Καταπολέμηση του εγκλήματος έχουν, έχει να κάνει συχνά με τα δικαιώματα του υπόπτου. Και σωστό είναι αυτό. Η ιδιωτική ζωή του υπόπτου, η σχέση του στη, στην ποινική δικονομία και στην ποινική δίκη καλή είναι. Αλλά την επόμενη πενταετία θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στη θέση των θυμάτων, ξέρετε. Και τα θεμελιώδη δικαιώματα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι απόλυτα. Κάθε φορά θα πρέπει να τα βλέπουμε και να τα ασκούμε σε ένα πλαίσιο. Όπως λέει και το Σύνταγμα στην Ολλανδία και αυτό ισχύει και για τους υπόπτους και για τα θύματα. Πρόεδρε, κατανοώ και συμφωνώ ότι το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή λέγει για τους τέσσερις φακέλους stop. Να περιμένουμε λίγο, μία πάυση για να περιμένουμε την 1η Δεκεμβρίου, τότε να έρθουν νέες προτάσεις και να δουλέψουμε ουσιαστικά με συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ραμόν Χαουρίγκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εδώ τώρα. Όλο το Κοινοβούλιο ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει ένα νέο νομοθετικό πακέτο για τα θέματα αυτά. Και ο κύριος Μπαρό καλοσυνάτος όπως πάντα, μας λέει ότι ερχόμαστε από μακριά. Έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό και πρώτη πρώτου του 2010 θα τεθεί σε ισχύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πρόβλημα. Εγώ κύριε Ντάλο, ε, Μπαρό, σας λέω από τώρα ότι θα πρέπει να ανακοινώσετε στο διάδοχό σας γιατί καταλαβαίνω ότι εσεί δεν μπορείτε να μας απαντήσετε για το μέλλον. Όταν θα έρθει εδώ στι ακροάσει στο Κοινοβούλιο, θα το ρωτήσουμε αν έχει την πρόθεση να κάνει νομοθετικό πακέτο για αυτό το ζήτημα. Γιατί το ζητάει σύσσωμο το Κοινοβούλιο. Και δεν είναι θέμα... Ε, ε, κάποιου νομοθετικού κνισμού. Δεν είναι ότι μας τρώει ε, στο Κοινοβούλιο για να επέμβουμε. Πρέπει να επέμβουμε. Γιατί έχουμε την νομοθετική αρμοδιότητα και εξουσία. Σε λίγες μέρες την αποκτούμε. Και αυτό το θέμα δεν είναι πια θέμα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εμείς θέλουμε να θεσπίσουμε ε, άλλο πλαίσιο, να κάνουμε άλλε προτάσεις. Παράδειγμα, εγώ σε πολλέ από τις οδηγίες ή σε πολλέ από τις αποφάσεις που έρχονται εδώ Βλέπω πολλές φορές πολλά ελλείμματα, πολλή νομική ανασφάλεια, ε, πολλά προβλήματα και εμείς θέλουμε να τα μεταρρυθμίσουμε. Πολύ ωραία να εργαστεί η Ευρωπόλ, ε, να εργάζεται και τώρα δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεχίσει, γιατί θέλω να προχωρήσει η Ευρωπόλα. Επίση, θέλω παρακαλώ να σεβαστείτε το δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Να μπορεί να έχει λόγο και να πει τι άποψη έχει για του κανόνε αυτού. Γιατί είναι νομοθετικό έργο και θέλουμε να το ασκήσουμε αυτό το νομοθετικό μα καθήκον. Γι' αυτό, όταν έρθει με το καλό επόμενο επίτροπο εδώ, θα το ρωτήσουμε και θα του ζητήσουμε να δεσμευτεί και να μα. Ε, υποσχεθεί ότι θα επιτρέψει το Κοινοβούλιο να νομοθετεί τίποτα παραπάνω. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Πεκ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω ένα στοιχείο επί της ουσίας και ένα επί της διαδικασίας. Η οικοδόμηση του χώρου ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας στην Ένωση είναι βεβαίως ε, επιταγή όλων αλλά είναι και να συνοδεύεται και από ένα μοντέλο δημοκρατίας που θα πρέπει να οικοδομήσουμε. Συμφωνούμε ότι η Ευρωπόλ θα πρέπει να προσαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά όλοι θέλουμε τα ανθρώπινα αλλά κυρίως τα τεχνικά μέσα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ε, των διαφόρων λαθερμπορίων να είναι αυστηρά οργανωμένο με ένα μέγιστο βαθμό νομικής ασφάλειας διότι εδώ αγγίζουμε την ίδια την καρδιά ε, των αρμοδιοτήτων μας, των εξουσιών μας που θα πρέπει να ασκούμε σε πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Στο όνομα της ομάδος μου θα ήθελα να πω στον κύριο Επίτροπο ότι όλη η δουλειά που έγινε δεν είναι καθόλου περιττή δεν είναι καθόλου μάταιοι. Θα ήταν όμως ακατανόητο και δεν θα μπορούσε ο Ευρωπαίος πολίτης να το δεχτεί Δηλαδή, ενώ περιμέναμε τόσο καιρό ε, την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας, τόσο καιρό επαναλαμβάνω, να μην έχουμε την υπομονή να περιμένουμε λίγες μέρες για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία με τη συνθήκη της Λισαβόνας να έχουμε δικαίωμα στην απόφαση στον τομέα. Είναι επίγον να περιμένουμε όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι επίγον να περιμένουμε και ως εκ τούτου και εγώ λυπούμε για την απουσία του Συμβουλίου διότι προς το Συμβούλιο κυρίως απευθυνόμεθα στο όνομα της Επιτροπής μου λοιπόν σας προτείνω να γίνει μια νέα νομοθετική πρόταση. Να περιμένουμε μια νέα νομοθετική πρόταση δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόμεβα ή Ρουέδα. Ο κύριος Ρούμε Ιρουδα. ευχαριστώ. Και εγώ στο όνομα των Πρασίνων θα ήθελα να λάβω τον λόγο για να επιμείνω ακριβώς επ' αυτού. Θα ήταν εντελώ ακατανόητο. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε τον ρόλο μας, περιμένοντας λίγες μέρες, να μην το κάνουμε. θα ήταν αδιανόητο και αδικαιολόγητο και έναντι του Ευρωπαίου πολίτη. Και κάτι άλλο τώρα για τα αστυνομικά εργαστήρια. Όταν μιλάμε για συντονισμό, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την αποκέντρωση. Από κοινού πάνε αυτά, χέρι-χέρι. Και το λέω γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει ένα εργαστήριο αστυνομικό, αλλά διάφορα, όπως στην Ισπανία. Mm. Είναι σημαντικό αυτό, να το γνωρίσουμε και να το διαδώσουμε ως πληροφορία, διότι δεν είναι ο συντονισμός μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά ο συντονισμός και σε επίπεδο κράτους μέλους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Βέρζια. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα επαναλάβω αυτά που είπαν ορισμένοι συνάδελφοί μου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατεπηγόντως πρέπει πριν από τη θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας να ασχοληθεί με την εφαρμογή τεσσάρων ε, κειμένων ε, για την προστασία της εμπιστευτικότητας δεδομένων που η Ευρωπόλ θα μπορούσε ε, να μεταδώσει και σε άλλα κράτη-μέλη ασχολούμεθα με κείμενα που είναι σημαντικά τα θέματα τους διότι θα, ε, θα... αρχίσουν να εμπίπτουν ε, στην συναπόφαση μετά την θέση εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Πολλοί θεωρούμε ότι οι συμπολίτες μας δικαιούνται ασφάλεια και ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μια προτεραιότητα όλα πρέπει να γίνουν ούτω ώστε οι συμπολίτε μας να μην ζουν συνεχώ με τον φόβο να είναι θύματα μια απόπειρα. Πρέπει όλα να γίνουν για να ενισχυθεί η αστυνομική συνεργασία. Αλλά αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει με οποιασδήποτε συνθήκες και όχι εις βάρος των θεμελιωδών δημοσίων ελευθεριών που είναι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στην ελευθερία κυκλοφορίας και ε, στην ελευθερία έκφρασης. Προσθέτω ότι η πρόληψη της εγκληματικότητας δεν γίνεται με μόνο περισσότερη ε, δίωξη ε, και καταπίεση θα πρέπει να προστατεύουμε τις ελευθερίες μας ως δημοκράτες και να τις καταστρατηγούμε μόνο σε απόλυτη ανάγκη. Η αστυνομική συνεργασία θα πρέπει να γίνεται σε ένα ε, ακριβές πλαίσιο νομικό που να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των ανταλλασσορμένων δεδομένων και την σωστή αναλογία των δεδομένων με τους στόχους ασφαλείας που έχουν τεθεί. Για το λόγο αυτό η ομάδα Γκουέντζελ ζητάει με άλλες ομάδες στο Συμβούλιο και στην Κομισιό να αποσύρει τις προτάσεις και εγώ λυπούμε που εδώ λείπει το Συμβούλιο από τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλοι. ο Πρόεδρος. Ο λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ. Αυτές οι εκθέσεις θέτουν τους κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, για την Ευρωπόλ ανάμεσα σε τα κράτη-μέλη και σε τρίτες χώρες ε, για ιδιωτικά δεδομένα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μη εγκεκριμένη ε, αποκάλυψη ορισμένων δεδομένων που δεν θα, που δεν θα πρέπει να θίγουν τα συμφέροντα της Ευρωπόλ. Τίποτα δεν γίνεται για την προστασία των, των πολιτών οι οποίοι φοβούνται μια τέτοια ανάγκη. Έχουμε επίσης ορισμένα δεδομένα για τις σεξουαλικές προτιμήσεις και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ε, έχουμε την Αλβανία, το Περού, την Ρωσική Ομοσπονδία, ε, η Ευρωπόλ. Ε, δεν νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι απαραίτητη, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να έχουμε την δική μας, το δική μας πολιτική δύναμη. οι επιφυλακτικοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουν ε, ότι υπάρχει ασελία από και προστασία για τα όσα κάνουν. Πολλοί που προέρχεστε από αστυνομικά κράτη, ίσως αυτό δεν έχει σημασία, αλλά ε, μια τέτοια για, τους, ε, για τις διοκτικές αρχές ε, είναι για το αγγλικό δίκαιο μια αντίληψη ξένη. Ενώ η Ευρώπη δημιουργεί δικαστικό σήμα όπως το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης την δίκη in absentia, εμείς στην Ευρώπη βλέπουμε πώς καταστρέφονται οι βασικές μας ελευθερίες με αυτόν τον τρόπο. Κάθε εισηγητής ε, τουλάχιστον είχε την εντιμότητα να πει ότι θα έπρεπε να απορριφθούν αυτές οι προτάσεις μέχρι ότου τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Αν είχε εντιμότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, θα επέτρεπε να τεθούν σε ισχύ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μάλτσερ, τελευταίος ομιλητής εξ ονόματος πολιτικών ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε τι κάνει η Ευρωπόλ. Δεν ε, είναι πάντα μεγάλη επιτυχία, αλλά πρόσφατα κατάφερε να ε, διαλύσει δίκτυα δουλεμπόρων και καταπολεμάει το διεθνές έγκλημα. Είναι καλό καταρχήν να υπάρχει συνεργασία διαφόρων αρχών για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Έρχομαι όμως τώρα στην προστασία των δεδομένων. Όταν είναι απεριόριστη η δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες όλων των αρχών, δεν εξασφαλίζεται η προστασία. Διαβιβάζονται σε διάφορες αρχές διάφορα στοιχεία χωρίς να υπάρχει καμία προστασία. Ακόμα και οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων στα διάφορα κράτη-μέλη πολύ γρήγορα γνωρίζουν όρια στη δράση τους και δεν μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά. Ούτε πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε κοινοτικό επίπεδο την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερο περιστέλλονται οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών στο βωμό της καταπολέμησης του εγκλήματος. Και τώρα έρχεται η Λισαβόνα. Το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης για τη συμφωνία των και την προστασία των χρηματικών συναλλαγών. Χρειάζονται ε, να προχωρήσουν γρήγορα και θέλουν όλοι να προχωρήσουν για το SWIFT και ξέρουν ότι δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Διότι αν δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές με το Σύνταγμα γιατί ε, να το δίνουμε χωρίς κανένα έλεγχο αυτό το δικαίωμα στην Ευρωπόλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όποιον άλλον θέλει. Όχι, δεν θα πρέπει να περάσει αυτή η ρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κύριε Μέλτσορ και τώρα ακολουθούν οι υπόλοιποι ομιλητέ. Όχι εξ ονόματος των ομάδων τους, ο καθένας προσωπικά. Ο κύριος Μπούσουτήλ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα γαλλικά και να τον ευχαριστήσω για το έργο του καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του που έχει την αρμοδιότητα αυτού του τομέα. Ελπίζω οι δύο πλέον επίτροποι, όχι ένας επίτροπος που θα τον διαδεχθούν να ε, μπορέσουν να εμπνευστούν από το πολιτικό σα όραμα, από την προσήλωσή σα και από το έργο σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Στα Μαλτέζικα τώρα. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε τώρα να μπω στην ουσία του θέματος. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ ε, το αρμόδιο γραφείο στη χώρα μου που ασχολείται με τα θέματα της Ευρωπόλ και τις σχέσεις ε, με την Ευρωπόλ και το όλο κλάδο του Σέγγεν. Στο γραφείο αυτό εργάζονται διάφοροι αστυνομικοί και φροντίζουν να συνεργάζονται αρμονικά και ταχαίως με άλλου ομολόγου του στα διάφορα κράτη-μέλη. Θέλω να του ευχαριστήσω και πραγματικά πρέπει να σα πω ότι κατά τη διάρκεια τη επίσκεψή μου εκεί κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η Ευρωπόλ. Κατανόησα πλήρω περί τίνος ε, πρόκειται και πόσο σημαντικό είναι να καταπολεμούμε την εγκληματικότητα. Ιδιαίτερα αυτούς τους καιρούς που ζούμε ε, ε, στην Ευρώπη που έχουμε ελευθερία στην κυκλοφορία. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε την πρόταση αυτή. Δεν είναι ότι έχουμε τίποτα με την Ευρωπόρ ούτε τίποτα εναντίον της. Αλλά θα θέλαμε να έχουμε λόγο κι εμείς ως κοινοβούλιο για την υπηρεσία αυτή που θα διαδεχθεί τώρα την Ευρωπόρ Για να είναι πραγματικά και πιο ισχυρή και να μπορεί να επομιστεί το έργο της σωστά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει για μισή λεπτό ο κύριος Κροτσέτα. Αγαπητέ αξιότιμε Πρόεδρε, συνάδελφε, η αίτηση εγκρίσεως του προγράμματος για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπόλ και άλλων εταίρων έχει ως εξής. Το σχέδιο, ε, αν ε, εγκριθεί, θα δημιουργήσει την σόλικη κατάσταση σύμφωνα με την οποία η ανταλλαγή πληροφοριών θα είναι δυνατή μεταξύ ευρωπολική και τρίτων χωρών χωρίς ακόμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει εγκρίνει τον κατάλογο αυτών των τρίτων. Το σχέδιο δίδει την εντύπωση όταν περιγράφει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ότι είναι μια αστήρευτη βάση δεδομένων που θα μπορούσε μάλιστα να τεθεί στη διάθεση τρίτων που το Κοινοβούλιο επιμένω δεν έχει ακόμα ορίσει. Το σχέδιο του Συμβουλίου, άρθρο 15 παράγραφος 2, λέει ότι σε περίπτωση ε, υπέρτατης ανάγκης και ανώτερης βίας μπορούν να μεταφερθούν δεδομένα για την ε, φιλοσοφική πίστη, για τη θρησκευτική πίστη, για την συνδικαλιστική δραστηριότητα και πολλά άλλα χωρίς ακόμα να ορίζεται αυτή η ανώτερη βία και η ίστατη ανάγκη. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον το Συμβούλιο να διευκρινίσει τι σημαίνει φιλή, τι σημαίνει εθνική ή εθνοτική προέλευση. Εμείς θεωρούμε ότι μία φιλή υπάρχει, η ανθρώπινη, που περιλαμβάνει γυναίκες και άνδρες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, διότι το πρόγραμμα, το σχέδιο αυτό του Συμβουλίου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ιδιαίτερα έτσι όπως παρουσιάστηκε ε, προσφάτως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρουτσέτα. Για ένα λεπτό τώρα Αλεξάνδρα Άλβανο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια του Σάιμον Μπουσουτήλ ε, για την εργασία του κυρίου Μπαρό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το έργο του και πολύ συχνά είχε τον άνεμο αντίθετα, αλλά να είστε βέβαιοι ότι εμεί η ομάδα των Φιλελευθέρων θα σα είχε δώσει μια ομπρέλα για να προστατευτείτε από τι καιρικέ αυτέ συνθήκε στη θύελα που διανύσατε συχνά. Μα φαίνονται περίεργα αυτά το που προτείνει το Συμβούλιο τώρα πριν την 30η Νοεμβρίου. Και βέβαια είναι φυσικό και επόμενο το Κοινοβούλιο να απορρίψει αυτέ τι προτάσει. Δεν σα φαίνεται κρίμα άλλωστε που δεν μας τιμάει με την παρουσία του και το Συμβούλιο για να τα ακούσει αυτά τα σχόλια. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα του διαβιβαστούν. Εγώ κανονικά ήθελα να μιλήσω για την έκθεση Κέρκοπ για τα εργαστήρια της επιστημονικής αστυνομίας και τις ε, προδιαγραφές και τα πρότυπα. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει να ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες ή να αρχίσουμε από εκεί να δούμε τι στοιχεία είναι αυτά που συλλέγουμε και πώς θα διαβιβάζουμε και αν θα πρέπει να διαβιβάζονται με το σωστό τρόπο. Γιατί πολλέ φορές βλάπτουμε τον ενδιαφερόμενο ότι να τον βοηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενο ομιλητής για 1,5 λεπτό είναι ο κύριο Στράσερ. Παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Μπαρό, σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και για την ε, κατανόηση ακριβώς τη σαφούς θέσεις του Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά τα διαδικαστικά. Εμείς δεν απορρίπτουμε τις προτάσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να τις διαμορφώσουμε. Αυτό είναι το αποφασιστικό που καθορίζει και την ψηφοφορία μας. Είναι σαφέστατο ότι η Ευρωπόλ είναι μία από τις επιτυχημένε ιστορίε που έχει να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του δουλεμπορίου, της ε, χρηματοδότησης, εγκληματικότητα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ε, η ευρωπαϊκή συνεργασία, η αστυνομική συνεργασία είναι πολύ σημαντική και είναι ακόμα σημαντικότερο να επεκταθεί και να εξαπλωθεί. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τη νέα βάση που δημιουργείται με τη νέα υπηρεσία, agency. Χρειαζόμαστε ανταλλαγή στοιχείων εδώ, χρειαζόμαστε συνδέσμους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Όλα αυτά τα χρειαζόμαστε ακριβώς για να συνεχίσουμε την ε, επιτυχημένη προσπάθεια και τη μάχη κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Τα ίδια όμως λόγια έτσι τόσο σταράτα θα πρέπει να τα λέμε και για την προστασία των πολιτών και των δικαιωμάτων τους. Εδώ έχουμε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, σαφείς ευρωπαϊκές αρχές και αξίες που καταγράφονται και στο ψήφισμα για το SWIFT, το οποίο περάσαμε το Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου μάλιστα, με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και αυτό που θα πρέπει να απαιτήσουμε από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η βασική γραμμή, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις τώρα με την Αμερική να επιβληθούν για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στράσερ. Και τώρα η κυρία Κίνγκα Γκέντς. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ που το Συμβούλιο ενδιαφέρεται για τη μετεξέλιξη και ανάπτυξη του δικτύου αυτού. Βέβαια κρίμα που απουσιάζει σήμερα το Συμβούλιο. Το είπαν και οι σε αυτό. Θα ήθελα να αφαιρθώ και στην ουσία και στη διαδικασία. Πριν από 10 χρόνια λήφθη απόφαση για το δίκτυο αυτό. Η αξιολόγηση τώρα έδειξε ότι το δίκτυο δεν εξύντλησε τις δυνατότητες που του δόθηκαν. Χρειάζεται ένα τέτοιο δίκτυο, χρειάζεται να αναπτυχθεί καλύτερα για να λειτουργεί καλύτερα. Η ε, κοινωνία των πολιτών, η συνεργασία ε, άλλους φορείς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, η πολιτική μας ομάδα ε, θεωρεί σημαντική τη λειτουργία και το έργο του δικτύου. Εμείς γιατί απορρίπτουμε αυτή την πρωτοβουλία. Σας εξηγήσαμε. Διότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το βήμα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής είναι ομιλήτρια η κυρία Βίκστρομ για ένα λεπτό, παρακαλώ största är att vi ännu inte har lyckats den ναι. ναι, δεν μπορεί κανείς να σταματήσει το εμπόριο των ανθρωπίνων όντων. Τα παιδιά και οι γυναίκες πολλούνται σαν εμπορεύματα ε, παντού στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ ήταν μισό εκατομμύριο γυναίκες που πουλήθηκαν στην Ευρώπη το 2009 πρέπει να μιλήσουμε για αυτές τις στρατηγικές τους ώστε να εξαλειφθεί αυτό το έγκλημα. Υπάρχουν όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πολεμούν το οργανωμένο έγκλημα και υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλά μειονεκτήματα σε αυτήν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, και του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής πρέπει να βελτιωθούν ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά εγκλήματα της ε, οργανωμένου εγκλήματος, της μαφίας ε, ε, και την, την, το εμπόριο των ανθρώπων. Σε λίγες μέρες θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά ίσως ε, ίσως θα πρέπει να ε, αναπνεύσουμε λίγο, διότι θα δούμε ότι θα είναι μια ευκαιρία ε, καλύτερης συνεργασίας, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Η Ευρωπόλ θα, θα αναβαθμιστεί, θα έχουμε καλύτερη συνεργασία με την Eurojust και θα μπορέσουμε να αναλάβουμε την καταπολέμηση του εγκλήματος στην Ευρώπη ε, εναντίον των συνδικάτων της μαφίας. Το 2009 νομίζουμε ότι δεν τιμά την Ευρώπη το εμπόριο των ανθρώπων για την εποχή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι σήμερα αυτή η συζήτηση και η συναφής απόφαση είναι μία πολιτική υφή συζήτηση. Βεβαίω. χρειαζόμαστε ενιαία πρότυπα αν θέλουμε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών και δικαστικών. Αλλά μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα σήμερα που είναι το πολύ σημαντικό ζήτημα που απορρέει από τη συνθήκη της Λισαβόνας η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων. Για να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Ως προς την νέα θέση ΠΕΚΣ πρόκειται για μια νέα θέση στην Ευρώπη που, από όπου απορρέουν πολλά ε, θετικά. Νομίζω ότι η νέα συμφωνία SWIFT θα περάσει από κόσκινο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τωρινά θέματα. Πριν ε, ε, την υπογραφή της συνθήκης Λισαβόνας ή μάλλον πριν την αρχή ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας εμείς αναρωτιόμαστε ε, γιατί ε, δεν θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε νέες προτάσεις και με αυτόν τον τρόπο το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάνουν την ευκαιρία να δώσουν εις ε, τους πολίτες Ευρώπης ένα θετικό σήμα για μια Ευρώπη των λαών. Πρέπει να απορρίψουμε αυτή την πρόταση γιατί θέλουμε να έχουμε μια πιο καλή συνεργασία συνεργασία και πρέπει να εφαρμόσουμε τώρα τα, ε, τις επιταγές και όχι αργότερα. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ορισμένα θέματα που αφορούν την ε, πρόληψη της, ε, του εγκλήματος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος. Θα πρέπει να δούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα σχετίζεται με την ανταλλαγή πληροφοριών και με πολιτισμικά δεδομένα. Ο Τζοβάνι Φαλκόνε διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο και αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα δράσει η Ευρώπη και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έπειτα το οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά ε, διαμέσου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα πολύ σοβαρά εγκλήματα. Δηλαδή τα εγκλήματα της μαφίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διότι η μαφία μπορεί να, η μαφία να διεισδύσει και, στα θεσμικά, και σε θεσμικά όργανα. Υπάρχει διαφθορά και αυτό το είδαμε και από πρόσφατες εκθέσεις το ελεγκτικό συνέδριο μίλησε και για ε, συγκεκριμένα εγκλήματα απάτης. Η κυρία Σαρατσάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Σκιώδης επί ενός ε, υποσκέλους της Europol δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτά που ήδη προελέχθησαν. Η Europol βοηθά τη διενέργεια έρευνων στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε στέναρα και να διευρύνουμε και τις αρμοδιότητες αυτού του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου θα εγκρίνει το φάκελο Europol χωρίς να αναμείνει την διαδικασία συναπόφασης που θα ισχύσει από 1η Άρα μιλάμε για ε, ένα νέο ευρωπαϊκό όργανο, τη Europol, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διευρυμένες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων της Europol, έτσι ώστε να μην υποσκάπτουν τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μόνικα Φλασίκο Μπαμπένοβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τομέας της ιατροδικαστικής έχει όλο και περισσότερο σημασία για την πάταξη των αξιοπίνων πράξεων και της εγκληματικότητα και μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα κοινό νομικό πλαίσιο που θα καθορίζεται η θέση όλων των ε, στοιχείων δηλαδή και των δικτύων και των εργαστηρίων και των ε, κανόνων συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, καμία κοινή κίνηση και αυτή η, αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Πρέπει δηλαδή το Συμβούλιο να εμπλακεί θα πρέπει να μπορέσει να υπάρχει ε, ένα πλαίσιο για την ε, για την έγκριση των διαφόρων ε, εργαστηρίων της της ιατροδικαστικής και δυστυχώς όμως παρόλο που έχουμε διατυπώσει προτάσεις σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν εισακουστεί. Ευχαριστώ. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία Catch the Eye. Ο πρώτος ομιλητής καλείται να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως νομικός και πρώην αστυνομικός θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου, η οποία στοχεύει όλα τα ιατροδικαστικά εργαστήρια τα οποία παρέχουν γενετικά δεδομένα να συμμορφώνονται με τον κανόνα 17025 που έχει σκοπό να ενισχύσει την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων ενώ αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο νομικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλήτης θα είναι ο κύριος Ζένσκα. Κύριε Ζένσκα παρακαλώ έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο. Εμείς επανερχόμαστε, θα επανέλθουμε αύριο σε αυτό το θέμα και κατόπιν θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, διότι αφενός θα θέλουμε να ενισχύσουμε ε, την αστυνομία και την Ευρωπόλ για να λειτουργούν αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά ωστόσο πρέπει να θυμούμαστε ότι εδώ παρεμβαίνουμε και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης και στον χώρο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Επειδή λοιπόν το θέμα αυτό δεν έχει λήξει, αφιστώ την προσοχή σας στο άρθρο 15 της απόφασης του Συμβουλίου που αναφέρεται στις, εκτελεστικές, στις διατάξεις εφαρμογής ε, των σχέσεων της Ευρωπόλ με τους εταίρους της και ειδικότερα για την ανταλλαγή δεδομένων. Μιλάμε για πολύ ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία πρέπει να ανταλλάσσονται μόνο αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Ποιο ωστόσο θα αποφασίζει ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη όχι. Αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye και θα παρακαλέσω τώρα τον Επίτροπο, τον κύριο Ζακ Μπαρό, να σχολιάσει αυτά που ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο το έργο μου. Ωστόσο θα ήθελα να αναφέρω ορισμένους λόγους οι οποίοι οδήγησαν την Επιτροπή σας να δεχθεί αυτή την παρουσίαση των κειμένων. Ας πάρουμε πρώτα το θέμα της Europol. Δύσκολα μπορούμε να διακόψουμε αυτή την μετατροπή του Europol σε υπηρεσία. Θα υπάρξουν βεβαίως και άλλα κείμενα και τότε θα συνομοθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει το έργο της Europol Και Άλλωστε στη διεύθυνση επικεφαλής της Europol αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος βρετανικής προέλευσης με πολύ μεγάλες ικανότητες. Θα ήταν λοιπόν λυπηρό να διακόψουμε κατά κάποιο τρόπο το έργο της προσπάθειας της Europol. Για τα άλλα δύο κείμενα θα ήθελα να πω ότι η διαπίστευση των εργαστηρίων, αναφέρομαι στο δεύτερο κείμενο, άλλα δύο κείμενα μάλλον για την διαπίστωση των εργαστηρίων είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλία του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Οπωσδήποτε είναι πρόοδο το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη έχουν δεχθεί την ιδέα αυτή τη διαπίστευση εργαστηρίων ώστε να έχουμε αξιόπιστα πλέον δεδομένα στη διάθεσή μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, μια πρόοδος. Τώρα, για τα δίκτυα. Εδώ δικαιολογούνται περισσότερο οι παρα, παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να το καθησυχάσουμε και να του δώσουμε νέες αποστολές στο μέλλον. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τον κύριο Στάθη και τον κύριο Μπουζουτήλ οι οποίοι παρατήρησαν πολύ σωστά ότι και ήταν και παρόν προηγουμένως ο πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ εγώ Είμαι πάρα πολύ προσιλωμένο στην ιδέα της ενεργού συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσα κατάφερα τα τελευταία χρόνια τα οφείλω στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πραγματικά λοιπόν, το γνωρίζετε άλλωστε, Επιθυμώ διακαώς τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θεωρεί ότι χρειάζεται μια εντελεχής κατά περίπτωση ανάλυση για να δούμε μήπως πρέπει να τροποποιήσουμε το κεκτημένο του τρίτου πυλώνα. Περάμε, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια μεταβατική ε, φάση. Περνάμε στην εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και είμαι βέβαιος ότι όλοι θέλετε να προωθήσετε μία συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικέ υπηρεσίες που θα σέβεται βεβαίως την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παρέμβαση του Κοινοβουλίου θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη ε, για αυτά τα μελλοντικά κείμενα και θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε περισσότερο την αστυνομική συνεργασία πάντοτε βεβαίως σύμφωνα με τις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με απόλυτο σεβασμό για τα δικαιώματα των πολιτών. Μιλάμε λοιπόν όμως για μια μεταβατική περίοδο ε, ε, αυτή τη στιγμή και αντιλαμβάνομαι την επιθυμία σας να συμμετάσχετε στην επεξεργασία αυτών των κειμένων αλλά η Επιτροπή μετά πιστεύω ότι με μια καταπερι... κατα... Ε, ε, ε, λεπτομερή ανάλυση κάθε περίπτωσης θα ξαναδούμε πιθανώς το κεκτημένο του τρίτου πυλώνα και αν έχουν ξεπεραστεί, απαρχιωθεί τα ισχύοντα κείμενα και χρειάζονται επικαιροποίηση ή τροποποίηση τότε θα διατυπώσουμε προτάσεις η διαδοχή μου ασφαλώς θα υποβάλουν προτάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν τότε στο Κοινοβούλιο να βελτιώσει τα κείμενα, τα νομικά, εφόσον πλέον θα συνομοθετεί. Και επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά ότι κύριε Πρόεδρε καθώς θα, ολοκληρώνω τη θητεία μου, θα λάβω σοβαρά υπόψη όλες οι υποδείξεις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε σαφώς επίγνωση του γεγονότος ότι θα προκύψουν πολλά νέα κείμενα για την αστυνομική συνεργασία και την δικαστική συνεργασία που θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν και να αναδιαμορφωθούν και σε αυτή τη διαδικασία θα υπολογίζουμε στην στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να τηρηθεί ως υπηρεσία η Europol, να συνεχίσει το έργο της και Παράλληλα θα σημειώσουμε τις ε, βελτιώσεις που θα επιφέρουν στο θέμα της διαπίστευσης των εργαστηρίων τα κράτη-μέλη και για την ε, ενίσχυση του δικτύου πρόληψης. Επαναλαμβάνω ότι αντιλαμβάνομαι τις θέσεις και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο μέτρο του δυνατού τις επόμενες εβδομάδες θα υπεραμεινθώ ε, αυτού του χώρου ελευθερίας και ισότητας που θέλουμε να χτίσουμε ως κράτη-μέλη με την υποστήριξη της συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα επόμενα λεπτά θα έχετε την ευκαιρία θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν το λόγο οι εισηγητές. Αρχίζουμε με τον κύριο Νίκολσον, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι απόψε είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση και θα ήθελα βέβαια εδώ να τονίσω ότι η Προεδρία έλαψε δια της απουσίας της Συμφωνώ απολύτως με τη Σόφιν Βέλτ. Βεβαίως θέλουμε να ενισχύσουμε μακροπρόθεσμα την Europol και να έχουμε μια συνεργάσιμη Europol. Πρέπει απλώς να δούμε τα οικονομικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, το οικονομικό έγκλημα, την τρομοκρατία τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά το ΕΛΚ ανέφερε ένα πολύ σοβαρό θέμα ε, συζήτησε τη θέση του θύματος σε σχέση με το δράστη και δυστυχώς βλέπουμε πάρα πολλές φορές και πολύ συχνά ότι αυτοί οι οποίοι είναι οι δράστες των εγκλημάτων ε, προσελκύουν μεγαλύτερη συμπάθεια από ότι τα θύματα. Έχουμε πολλούς τομείς όπου μπορούμε αυτό να το αποδείξουμε και δεν είναι δυνατόν αυτό να θεωρηθεί σαν κάτι το αποδεκτό διότι πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε όλο και περισσότερη βοήθεια στα θύματα διότι δεν είναι δυνατόν ο δράστης του εγκλήματος να έχει ίση μεταχείριση με το θύμα δεν μπορεί όμως κάτι τέτοιο να γίνει χωρίς συνεργασία και αυτή είναι η πραγματικότητα ατυχώς. Γι' αυτό και ε, θα πρέπει να δούμε ότι ε, τελευταίως ε, διαπιστώσαμε στην Αγγλία συνεργασία μεταξύ των αρχών της Βορείου Ιρλανδίας και των Βρετανικών αρχών και μπόρεσαν να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι διακινούσαν εκατομμύρια τσιγάρα. Άρα χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται πιο ισχυρή Europol και θα πρέπει να, όλοι να συνεργαστούμε προς όφελος όλων μας. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Βέλτ. Πριν κάνω την παρέμβασή μου, θα ήθελα και εγώ να ε, εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Επίτροπο Μπαρό και να του πω ότι θέσατε πολύ υψηλές προδιαγραφές για αυτόν που θα αναλάβει στη συνέχεια το έργο σας. Δεν θα μπω στο περιεχόμενο, αλλά στη διαδικασία, γιατί θα ήθελα να διασαφηνίσω το εξής. Άκουσα έμεσα από το κενό έδρανο εκεί απέναντι ότι υπάρχει πολύ καλός λόγος, ε, που, πολύ μεγάλη σκοπιμότητα που επιταχύνει τη διαδικασία το Συμβούλιο, διότι η Europol πρέπει να γίνει θεσμικό όργανο μέχρι την πρώτη Πρώτου. Αν όμως το Συμβούλιο ε, ασχολιόταν πραγματικά με τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να είναι παρόν, να είχε αρχίσει τις διαδικασίες πριν από τα τέλη Ιουλίου και να δεχτεί την προσφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τάχιστη διαδικασία, διότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη σοβαρά τις ευθύνες του και εργαζόμαστε με μεγάλη σπουδή εκεί που πρέπει. Προτείνουμε αυτή τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο που διέπεται από το πνεύμα της Λισαβόνα. Ζητήσαμε ε, ε, επέκταση κατά ένα μήνα, αλλά δεν μας το χορήγησε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έλαμψε δια της απουσίας του σήμερα και αυτό καταδεικνύει ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και λυπάμαι ιδιαίτερα γι' αυτό, διότι ε, βρισκόμαστε 7 μέρες πριν από το στόχο μας. Πρέπει να συνεργαστούμε και θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για εγωιστικά κίνητρα για το εγώ μας, ούτε για το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε για τα εθνικά κοινοβούλια που προβάλλουν τον εαυτό τους. Μιλάμε για, για το ότι είμαστε υπόλογοι έναντι του κοινού. Μιλάμε δηλαδή για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, δηλαδή ε, στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα των πολιτών μας και υπόλογο είναι το Συμβούλιο, πολύ περισσότερο από εμάς. Άκουσα αυτά που μας είπε ο Επίτροπος, θα ήθελα όμως μία δήλωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εφόσον δηλαδή πρόθεσαν εντάχει το όλο πακέτο υποσχέθηκαν ότι θα αποσύρουν ή θα αναθεωρήσουν την απόφαση το ταχύτερο δυνατόν. Το αργότερο μέσα σε έξι μήνες και μετά θα συμμετάσχει ενεργά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης, διότι είμαστε και εμείς υπόλογοι έναντι των πολιτών. Ο κύριος Άλμπρεχτ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εργασία που έχει κάνει σε σχέση με την Ευρωπόλ και να σας πω ότι το θέμα δεν είναι εδώ η ε, Ευρωπόλ να ε, μετατραπεί σε ένα ε, γραφείο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να εμποδιστεί. Το θέμα είναι οι αρμοδιότητες και είναι πολλοί οι οποίες θα τις ανατεθούν και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και θα πρέπει να συζητήσουμε συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξοδικά για να μπορέσει να έχει νομιμοποιηθεί. Όπως άλλωστε ρέχλη βλέπουμε ότι το Συμβούλιο δεν παρίσταται καν για να ακούσει αυτή την κριτική η οποία είναι ουσιώδης για μια δημοκρατία. Ελπίζω λοιπόν τώρα ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να ακολουθήσει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία. Χρειαζόμαστε Είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική συζήτηση και για ε, τα μέτρα αλλά και για την αποτελεσματικότητά τους και εκεί θα πρέπει να ενισχυθούν και να συμμετάσχουν περισσότερο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ τον εισηγητή που παρουσίασε αυτές τις απαιτήσει και θα ήθελα και το Συμβούλιο να μπορέσει να συμπεριφερθεί αναλόγως και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Δίας Ντεμεράε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ υποστηρίζω τη Europol και θα ήθελα το συντομότερο δυνατόν να διαθέτει όλα τα κατάλληλα μέσα, έμψυχο υλικό και πόρους για να φτάσει στους απότερους στόχους της. Όπως ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνα, Συνοψίζοντας, τι είναι η Europol, σε τι συνίσταται. Δεν είναι διακυβερνητική, διακυβερνητικός φορέας, είναι θεσμικός, ενδοκινοτικός φορέας, αλλά είναι ένας ευάλωτος φορέας τη στιγμή που δεν υπόκειται σε πλήρη έγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη σπουδή έτσι ώστε να περιοριστεί ο έλεγχος του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η βασική αρχή. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχτούμε το Συμβούλιο να κινείται με αυτό τον τρόπο θελοτυφλίας. Χρειάζεται μία δήλωση, μία σαφής δήλωση, έτσι ώστε να υποβληθεί ένα νομοθετικό πακέτο πριν από έξι μήνες, όπως ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό που επιπλήττουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε έξι εκθέσεις σε μια μισή ώρα ως προς θέματα ύψης της σημασίας, γιατί μιλάμε για την πρόληψη του εγκλήματος, μιλάμε για τα εργαστήρια ανακριτικής και για τέσσερις εκθέσεις ως προς το ρόλο της Europol. Ξέρουμε τη σημασία της συζήτησης, αλλά το σώμα δεν μας επέτρεψε να εμβαθύνουμε το όλο θέμα μέσα σε μια μισή ώρα. Δεν μπορούμε να συζητάμε έξι εκθέσεις σε μια μισή ώρα. Θα πρέπει να είμαστε πιο ορθολογιστές μελλοντικά έτσι ώστε τέτοιες σημαντικές συζητήσεις να μας απασχολούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αύριο θα ε, αποτανθούμε στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δίας Ντεμέρ. Η ε, κυρία Αλφάνο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μπάρο διότι συμμερίστηκε τις ανησυχίες μας εμείς ε, δεν θέλαμε να πούμε ένα απλό όχι στο Συμβούλιο, αλλά επειδή σε λίγες μέρες θα μας διέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, νομίζω ότι ο ρόλος της συναπόφασης του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός. Ζήτησα από το Συμβούλιο να προτείνει αμέσως μετά τη Λισαβόνα μία πρόταση πολύ πιο φιλόδοξη σε σχέση με το δίκτυο πρόληψης εγκλήματος. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό χρειάστηκε να απορρίψουμε το όλο πλαίσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να δρά με συναπόφαση σε τόσο σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ την κυρία Νίκολσον γιατί μίλησε για τα θύματα, το ρόλο των θυμάτων και τις μεγάλες σφαγές που έχουν γίνει. Πολλές φορές αντιστρέφονται οι ρόλοι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταπολεμήσαμε την τρομοκρατία, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε τόσο ε, έντονα το οργανωμένο έγκλημα. Δεν μπορούμε παρά να λάβουμε υπόψη ένα μεγαλύτερο δίκτυο πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτά που ο κύριος σε σχέση με αυτά που είχε πει ο δικαστής Φαλκόνε που σκοτώθηκε από τη μαφία. Πολύ συχνά. Γίνεται σύγχυση μεταξύ ε, θύματος και σφαγέων και υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν το προσέχουν αυτό. Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες ε, εντάσσουν τα θύματα της ε, τρομοκρατίας και τα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια τυπολογία. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, διότι τη στιγμή που μιλάμε για μια καινοτόμο πολιτική, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ομοιόμορφη αντιμετώπιση. Ευχαριστούμε. Έχει λήξει η κοινή συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Ζακ Μπαρό για την ε, ιδιαίτερα υπεύθυνη, τον ιδιαίτερα υπεύθυνο ρόλο του. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη,